items on our agenda still. So, let's Δύο πράγματα έχουμε ακόμα στην ημερήσια διάταξη, συνάδελφοι. Προχωράμε λοιπόν. 16 ως 20 κοινή συζήτηση για την Συμφωνία Ελευθερου Εμπορίου με την Σιγκαπούρη. Η συμφωνία ίδια και το κομμάτι προστασίας των επενδύσεων. Να τα συζητήσουμε αυτό μαζί. ήθελα πρώτα απ' όλα να καλωσορίσω την κυρία Ρούσο που συνέταξε την μελέτη, την κυρία Ρούσο που συνέταξε την μελέτη. Καλώς ήρθατε και έχουμε και κάποιους προσκεκλημένους από την Σιγκαπούρη που ελπίζω να έρθουν σύντομα.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 και η προσκεκλημένη από την Σιγκαπούρη, ο Υφυπουργό Εμπορίου, κάθεται δίπλα μου, ο κύριος Λουκ Γκο, ο πρέσβης, ο κύριος Ράτναμ και εκπρόσωπος των ε, Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων στην Σιγκαπούρη, η κυρία Κορνέλης, που κάθεται εκεί μάλιστα. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω και Έχουμε μία ώρα για την συζήτηση της ε, συμφωνίας και της μελέτης. Και θα προσκαλέσω. Θα δώσω τώρα τον λόγο στην κυρία Ρούσου για να μας δώσει μια γενική εικόνα για την μελέτη ε, για στα πέντε λεπτά. Ευχαριστώ. Η μελέτη προβλέπει μια συνολική ανάλυση των διατάξεων της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου με την Σιγκαπούρη και χωρίζεται σε πέντε σκέλη. Το πρώτο περιγράφει το πεδίο εφαρμογής συμφωνίας, δηλαδή το μίσο πίσω απελευθερώνεται η πρόσβαση στην αγορά με τη μείωση παραδείγματος χάρη των δασμών ή τη μείωση των μη δασμολογικών εμπορίων. Το δεύτερο τμήμα κοιτάει ζητήματα της νέας γενιάς ε, εμπορικών συμφωνιών όπως η προστασία των επενδύσεων και η πνευματική ιδιοκτησία και τα συγκρίνει με άλλες συμφωνίες νέας γενιάς που διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να σημειώσουμε ότι το επενδυτικό κεφάλαιο που αξιολογήσαμε ήταν το κείμενο του Μαΐου 2015 καθώς η αναθεωρημένη συμφωνία δεν ήταν τότε διαθέσιμη. Το τρίτο σκέλος της ε, μελέτης ε, κάνει μία πρόβλεψη για τον πιθανό αντίκτυπο της συμφωνίας ε, στις οικονομίες Σιγκαπούρης και Ευρωπαϊκής Ένωσης και κοιτά ακριβώς τις αντιδράσεις των ενδιαφέρουμενων μερών. Ένα τέταρτο σκέλος κάνει μία ανάλυση της απόφασης του δικαστηρίου στην υπόθεση 2 15 για την ε, υπογραφή των, της συμφωνίας από τα κράτη-μέλη και τις συνέπειες αυτής της απόφασης και τέλος έχουμε κάποιες ε, συστάσεις και συμπεράσματα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας βλέπουμε ότι οι, προβλε... οι πρόνοιες της ε, συμφωνίας θα, θα σημάνουν απελευθερωμένο εμπόριο σε μεγάλο βαθμό. Βεβαίως ε, δεν μιλάμε σε τόσο μεγάλο βαθμό όπως σε άλλες περιπτώσεις καθώς η Σιγκαπούρη de facto έχει μηδενικούς δασμούς οι εξαγωγοί στη Σιγκαπούρη θα μπορούν τώρα να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά επιπλέον ε, θα διευκολυνθεί και το εμπόριο στις υπηρεσίες, ε, κάτι το οποίο θα είναι σημαντικό και για τις δύο πλευρές, δεδομένου του ότι η Σιγκαπούρη είναι σημαντικός κόμβος παροχής υπηρεσιών. Στην σύγκρισή μας των διατάξεων των, νέων, της, των συμφωνιών της νέας γενιάς, συγκεκριμένα με την ΣΥΤΑ και την συμφωνία με την ε, Κορέα, βλέπουμε ότι η νέα αυτή συμφωνία είναι συμβατή με τη νέα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όσον αφορά την προστασία των επενδύσεων. Το κείμενο της νέας το οποίο εξετάσαμε για τους σκοπούς αυτής της παρουσίασης, είναι πολύ πιο κοντά ε, με αυτό της ε, ΣΥΤΑ από το αρχικό κεφάλαιο επενδύσεων. Παραδείγματο χάρη καθορίζει ένα μόνιμο δικαστήριο και ε, μια διαδικασία εφέσεων. Όμως οι διαφορές μεταξύ των δύο κειμένων θα μπορούσαν να αποδειχθούν σημαντικές στην πράξη, όπως παραδείγματο χάρη το πεδίο εφαρμογή της ρήτρα μη διακριτικής μεταχείρισης. Και μετά από συνεντεύξεις βλέπουμε πως οι αντιδράσεις είναι γενικά θετικές, καθώς αυτοί οι οποίοι μας απάντησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Σιγκαπούρη θεωρούν ότι η συμφωνία είναι φιλόδοξη και θα προσφέρει νέες ευκαιρίες για εμπόριο και επενδύσεις και θα δημιουργήσει θέσει εργασία. Όμως, εκφράστηκαν κάποιες ανησυχίες. Ιδιαίτερα εκπρόσωποι των Συνδικάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασαν ανησυχίες για την έλλειψη ενός μηχανισμού κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης ε, των εργατικών δικαιωμάτων, καθώς και την γενικότερη μη εφαρμοσμούτα του κεφαλαίου για την βιώσιμη ανάπτυξη. Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι οι Σιγκαπούροι δεν είχαν αυτές τις ανησυχίες και είπαν ότι η Σιγκαπούροι επιβάλλει υψηλές προδιαγραφές ε, προστασίας ε, των εργαζομένων οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι εξέφρασαν την δυσαρέσκειά τους με τη μεγάλη καθυστέρηση στην διαδικασία κύρωσης. Στην ε, σύνοψή μας της απόφασης του δικαστηρίου 2 κάθετος 15 ε, βλέπουμε ότι κατά την άποψη του δικαστηρίου υπάρχουν δύο πτυχές στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κοινή αρμοδιότητα με τα κράτη-μέλη. Η πρώτη πτυχή είναι επενδύσεις που δεν θεωρούνται άμεσες ξένες επενδύσεις και η δεύτερη πτυχή είναι ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών. Η συνέπεια αυτής της απόφασης είναι ότι είναι πολύ πιθανό τα μελλοντικά κεφάλαια να απαιτήσουν την έγκριση όλων των κρατών μελών. Όμως, η ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και των κρατών μελών να συνάψουν τέτοιες συμβάσεις οι οποίες θα περιέχουν έναν μηχανισμό επίλυσης διαφορών που θα αφαιρούσε την δικαιοδοσία αυτή από την αποκλειστική αρμοδιότητα του δικαστηρίου πλέον τίθεται ένα αμφιβόλο και άρα θα μπορούσε το ζήτημα να γίνει πλέον καθαρά ακαδημαϊκό. Θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο στον συναδελφό μου, τον κύριο Κλίν Τζέιμπερς από την Capital Economics, ο οποίος επίσης θα ήθελε να πει δύο λόγια. Θα αναφερθώ εγώ στην οικονομική πτυχή εξετάσαμε την μελέτη στο εμπόριο, στις επενδύσεις και στην οικονομία γενικότερα, ξεκινώντας από το εμπόριο. Σε γενικές γραμμές η επιστημονική έρευνα λέει ότι το ε, ελεύθερο εμπόριο είναι υποφελές και για τις δύο πλευρές ε, και τα ωφέλη είναι αρκετά μεγάλα. Εξετάζοντας την ε, Κορέα που είναι η πιο παρόμοια συμφωνία με αυτήν, βλέπουμε ότι υπήρξε οπωσδήποτε αύξηση των εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Νότια Κορέα από όταν ετέθη αυτή η συμφωνία εν ισχύ και η κατάσταση ήταν κάπως πιο δύσκολη όσον αφορά τις εξαγωγές της Νότιας Κορέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες μπορεί και να έπεσαν μάλιστα την περίοδο που εξετάζουμε αλλά αυτό μάλλον δεν οφείλεται στην συμφωνία αλλά οπωσδήποτε θα υπάρχουν ωφέλη για τους νότιοκορεάτες καταναλωτές όσον αφορά τις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης το κοιτάξαμε από την οικονομετρική σκοπιά για να δούμε διαφορά άλλα ζητήματα όπως εποχιακά αποτελέσματα και τις ε, υπάρχουσες τάσεις και βλέπουμε ότι οπωσδήποτε υπήρχε κάποιο αποτέλεσμα για τις εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ένωσης. Ε. Όμως βεβαίως η συμφωνία αυτή διαφέρει όσον αφορά το περιεχόμενο και την αφετηρία των ε, οικονομιών και του εμπορίου οπωσδήποτε. Τέλος, ε, η συμφωνία που υπέγραψε η Σιγκαπούρη με την Κίνα φαίνεται ότι τα επόμενα χρόνια κατέληξε σε μία μείωση των εισαγωγών ε, από Νότια Κορέα και είπα στην Σιγκαπούρη. Οπότε κοιτώντας μετά τον αντίκτυπο για την ε, Σιγκαπούρη φαίνεται ότι η αύξηση θα είναι μικρότερη από ό,τι στην περίπτωση της ε, Κορέας και αυτό γιατί η μεταβολή στους δασμούς είναι σαφώς μικρότερη. Ήδη η Σιγκαπούρη προσφέρει πρόσβαση χωρίς δασμούς. Παρόλα αυτά θα υπάρξει μια άρση των μη δασμολογικών φραγμών και για τις εξαγωγές της Σιγκαπούρης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει το αντίθετο. Σε αντίθεση με την Κορέα θα έχουν μεγαλύτερη μείωση των δασμών και όσον αφορά τους κανόνες προέλευσης, οπότε υπολογίζουμε ότι και οι δύο πλευρές θα αυξήσουν τις εξαγωγές τους κατά 10% όσον αφορά τις επενδύσεις. Και πάλι οι γενικές μελέτες δείχνουν ότι οι συμφωνίες ελευθερίου εμπορίου έχουν γενικά ευεργετικό αποτέλεσμα και επίδραση στις επενδύσεις. Υπήρχε σημαντικός αντίκτυπος από την Κορεατική Συμφωνία και στην περίπτωση της συγκεκριμένης αυτής ε, συμφωνίας υπάρχουν κάποιες επιπλέον πτυχές ε, όπως ένας μηχανισμός επίλυσης ε, διαφορών αν και ακόμα δεν έχει αποφασιστεί κάτι τέτοιο αλλά συνολικά αναμένουμε ότι θα αυξηθούν οι επενδύσεις όπως έγινε με την Κόρεα και θα υπάρχει άρα μια αναλογική αύξηση και για τις δύο πλευρές και τέλος κάναμε μια συνολική μακροοικονομική αξιολόγηση με συγχωρείτε δεν ξέρω αν έχω ξεπεράσει τον χρόνο μου. Το βλέπετε εδώ, έχουμε βάλει και το εμπόριο και τις επενδύσεις για το συνολικό αποτέλεσμα στο ΑΕΠ. Υπάρχουν μελέτες που μετράνε ε, το πώς ακριβώς ε, έχει αντίκτυπο η αύξηση του εμπορίου και των επενδύσεων στο ΑΕΠ. Ε, θα υπάρχουν λοιπόν μικρή, αλλά... μικρά αλλά θετικά αποτελέσματα και στις δύο οικονομίες. Σας ευχαριστώ. Ποιος θέλει τώρα να σχολιάσει. Θα δώσω πρώτα το λόγο μάλλον στον ε, κύριο Γκουένο για να σχολιάσει την ε, άποψη της ε, Σιγκαπούρης και πρώτα ο Ντέιβιντ Μάρτιν. Ευχαριστώ που είναι ο εισηγητή. Όπω γνωρίζουν οι συνάδελφοι, αυτή η συμφωνία είναι τόσο παλιά, όπου η Βρετανία είχε μια αίσθηση κυβέρνηση όταν ξεκινήσαμε αυτή τη διαπραγμάτευση. Τώρα είμαστε σε τελείω διαφορετικέ περιστάσει. Δεν είναι προφανώ η πρώτη συζήτηση για την συμφωνία με τη Σιγκαπούρη, αλλά είναι η πρώτη που κάνουμε. Δεν θα να ανατρέξω το ιστορικό γιατί το γνωρίζετε πήγαμε στο δικαστήριο και άλλη δικαθυστέρηση επειδή χωρίσαμε τις δύο συμφωνίες και ούτε καθεξής θέλω να πω εξ αρχής ώστε να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ως εισηγητής υποστηρίζω απόλυτα την ολοκλήρωση αυτών των συμφωνιών είναι καλές για τη Σιγκαπούρη και για την Ένωση πιστεύω να εξηγήσω καταρχάς γιατί ε, είμαι αυτή της άποψης όσον αφορά την ε, Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου υπάρχουν ωφέλη, είναι ασφαλές κράτος Σιγκαπούρη και χρησιμεύει ως κόμβος για ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη και όσο περισσότερο εμπόριο έχουμε με τη Σιγκαπούρη σημαίνει τόσο περισσότερο εμπόριο έχουμε με ολόκληρη αυτή την περιοχή. Έχουμε πάνω από 10.000 ευρωπαϊκές εταιρείε που κρατούν γραφεία στη Σιγκαπούρη και πολλές εξ αυτών έχουν και το περιφερειακό τους επιτελείο στη Σιγκαπούρη. δεν αναμένουμε να καταργηθούν όλοι οι δεσμοί από την πρώτη μέρα, αλλά υπάρχει πρόβλεψη για σταδιακή μείωση, θα υπάρξουν καλύτερες ευκαιρίες για τους Ευρωπαίους επιχειρηματίες και ως προς αυτό να τονίσουμε ότι χρησιμοποιείται ένα θετικό κατάλογος για τις υπηρεσίες σύμφωνα με το πρότυπο GATT. Για πολλούς συναδέλφους, αλλά ιδιαίτερα για τους Ιταλούς συναδέλφους, φαντάζομαι, θα εγγυηθούμε την ε, ε, διατήρηση πάνω από 200, 200 GIE από τη στιγμή που έχει επικυρωθεί η συμφωνία. Πρέπει να πούμε πως πρόκειται για μια προοδευτική εμπορική συμφωνία όπου πολλές από τις αξίες τις οποίες μας είναι ιδιαίτερα προσφυλείς στηρίζονται. Δεν θα οδηγήσει σε μείωση των προτύπων μας. Ε, τα αγαθά που προέρχονται από τη Σιγκαπούρ θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα ε, στάνταρ της Ένωσης. Ε, θα υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, Βλέπετε η αρχή της προφύλαξης, διαχείριση περιβάλλοντος, διαχείριση αλληλείας και δασοκομεία. και Βεβαίως συμπεριλαμβάνονται οι στάνταρ δεσμεύσεις για τα εργατικά δικαιώματα, τις συμβάσεις ε, του Διεθνούς ε, Γραφείου Εργασίας και όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα η, η Σιγκαπούρη θεωρείται ε, ο παράδεισος της Νοτιοανατολικής Ασίας αν δει δηλαδή κανείς τι συμβαίνει δίπλα. Ωστόσο πρέπει να γίνουν κάποιες βελτιώσεις ακόμα. Η Σιγκαπούρη πρόσφατα έχει συνεργαστεί με το Διεθνές Γραφείο εργασία. Έχουμε επισκεφθεί μαζί την χώρα για να συζητήσουμε πώς μπορούν να γίνουν περαιτέρω προσπάθειες για την ε, ε, κύρωση άλλων συμβάσεων του Γραφείου Εργασίας. Δεν προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων, αλλά σε περιπτώσεις παράβασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουμε ρήτρα ασφαλείας που μας επιτρέπει να αναστείλουμε και τις δύο συμφωνίες. Τροποποίησεις μπορούν να γίνουν μέσω της ε, γενικής ρήτρα αναθεώρησης και, και δεν κάνουμε ε, υποσχέσεις η Σιγκαπούρη είναι ανοιχτή για διαπραγματεύσεις για αυτά τα θέματα. Και αν δει κανεί την παγκόσμια κατάσταση, η συμφωνία θα είναι η πρώτη εμπορική συμφωνία που θα συναυθεί ανάμεσα στην Ένωση και μια ασιατική χώρα. Όπως γνωρίζετε, είναι ένας ε, στόχος ε, να συναυθεί μια περιφερειακή εμπορική συμφωνία εγώ γι' αυτό ήμουν ε, ε, εισηγητής για πολλές διμερείς συμφωνίες στην Ασία. Ακόμα δεν έχει κυρωθεί καμιά άλλη. Συναγωνιζόμαστε. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην μείνει πίσω ενώ οι εμπορικοί μας εταίροι προχωρούν προς ε, εντατικότερες εμπορικές ροές. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε πια στις ΗΠΑ, γι' αυτό η ενίσχυση των σχέσεων μας με την Νότια Ανατολική Ασία είναι επίγουσα και πάλι η Σιγκαπούρη είναι, και μάλλον η Νότια Ανατολική Ασία είναι μια από τις περιοχές του κόσμου που αναπτύσσονται όσο ε, γίνεται ρηγορότερα, ταχύτερα. Τώρα, για την ε, IPA, όπως ανέφερα και πριν, για τις, ε, την προστασία των επενδύσεων θέλουμε να αντικαταστήσουμε το ISTS με το σύστημα ε, προστατευμένων επενδύσεων και θυμίζω ότι το Κοινοβούλιο ήταν κατά του ISDS, του συστήματος για ε, τη διευθέτηση των διαφορών μεταξύ κράτους και επενδυτή. Ζητήσαμε να δημιουργηθεί ένα μόνιμο δικαστήριο ένα κώδικα διδολογίας για τους δικαστές ώστε να αποφευθούν οι συγκρούσει συμφερόντων και να εξασφαλίσουμε την και συμπεριφορά, δημοσίευση και των βασικών ε, κειμένων ε, online, καθώς και προσπάθεια για ένα ε, σύστημα θέσπισης, μάλλον για τη θέσπιση ενός συστήματος πολυμερούς δικαστικού συστήματος. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στη συμφωνία. Όλα όσα ζητήσαμε λοιπόν είναι μέσα στη συμφωνία. Οπότε κατά τη γνώμη μου οι διατάξεις για την προστασία των επενδύσεων ξεπερνούν και τα όσα επιθυμούσαμε. Ε, είναι και στην συμφωνία ΣΕΤΑ ε, Έχουμε λοιπόν ε, ε, την θέσπιση ενός ε, δικαστηρίου για τη διευθέτηση των διαφορών, κώδικα δεντολογίας, διορισμό, προβλέπεται ο διορισμός, ο μελλοντικός διορισμός των δικαστών σε περίπτωση που κάποιο μέλος του δικαστηρίου εγκαταλείψει τη θέση του, παραιτηθεί οτιδήποτε και όλα είναι, προβλέπεται να είναι πιο προσβάσιμα για τις μικρομεσαίες. Πολλά από αυτά που ζητήσαμε στην ΣΕΤΑ υπάρχουν και πολλά ωφέλη, είναι και περισσότερα. Θα ήταν παράξενο να ζητάμε ένα πολυμερές σύστημα και να μην στηρίξουμε το πρώτο, την πρώτη συμφωνία που περιλαμβάνει αυτά τα συστήματα που εμείς ζητήσαμε. Γι' αυτό και σας συστήνω να εγκρίνουμε αυτές τις δύο συμφωνίες. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κ. Γκόγια, πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Μάρτιν, ε, για την ευκαιρία που μας δίνεις να συζητήσουμε αυτές τις δύο συμφωνίες, οι οποίες δεν είναι καινούριε. Ε, και θα ήθελα να επισημάνω κάποια σημεία ε, που είναι σημαντικά όσο συζητούμε τη δικασία κύρωσης. Τα σημεία αυτά είναι το πώς ε, θα πρέπει οι συμφωνίες αυτές να ενταχθούν σε ένα διεθνές ε, πλαίσιο. Η κάθε περιφέρεια έχει κάποιες ε, ευκαιρίες τρίτων, ειδικέ εισφορές και θέματα τα οποία, με τα οποία ασχολούνται οι δύο αυτές συνθήκες. Είναι σημαντικά θέματα, η διαφάνεια, το περιβάλλον, που, για παράδειγμα που υποφελούν και τις δύο πλευρές των ε, συμφωνιών. Ε, ε, βεβαίως υπάρχουν ε, διάφοροι γενικευμένοι δασμοί που δημιουργούν προβλήματα στο χάλιβα κλπ τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η Σιγκαπούρη κάνουμε το καλύτερο δυνατό τους ώστε να επιληθούν τα προβλήματα αυτά και ταυτόχρονα είμαστε ευαισθητοποιημένοι όσον αφορά την υποστήριξη του διεθνούς ε, πλαισίου, όσον αφορά και την πρόοδο των υποχρεώσεων για το περιβάλλον. Ε, ε, θα πρέπει να υπάρξει ένα χειρό μήνυμα εκ μέρους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σιγκαπούρη ότι θέλουμε να προχωρήσουμε στη σύσταση θέσεων απασχόληση και να στηρίξουμε το διεθνές πλαίσιο ενθαρρύνοντας ε, για παράδειγμα τη ε, ε, σχέση με την Ιαπωνία μαζί με τον ΠΟΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε σε όλες αυτές τις πλατφόρμες Πολλές, ε, πολλές από τις διασυνδέσεις που δημιουργήσαμε ε, ε, μέχρι στιγμή στο Μεξικό και η Ιαπωνία έχουν ήδη κυρώσει τη συμφωνία και υπάρχει στην περιοχή αυτή της Ανατολικής Ασίας και υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες θα προχωρήσουν στην υπογραφή, στην κύρωση συμφωνίας είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα της διασύνδεσης με την Ασία, με την Ανατολική Ασία. Ε, εν ολίγης ε, υπάρχει μεγάλη σημασία στην υπογραφή αυτής της ε, συμφωνίας για όλους τους ενεχόμενους φορείς, όχι μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά και για τους εργαζόμενους σε σχέση με τις προδιαγραφές, με τα πρότυπα εργασίες, ε, που θα πρέπει να γίνονται σεβαστά και δεν θα πρέπει να, δεν θα πρέπει να αποφασίζονται μερός. Τώρα, το δεύτερο ε, σημείο ε, μπορείτε να δείτε στα δεδομένα τα οποία έχουμε στην Σιγκαπούρη έχει υπάρξει δυνατότητα για πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αποκτήσουν μια πρόσβαση στην ε, περιοχή αυτή και στη Μαλαισία κλπ. Ε, ε, είναι μια τεράστια οικονομία αυτή τη στιγμή. θα συνεχίσουμε να διευκολύνουμε τα αποτελέσματα αυτά και να δημιουργήσουμε μια γέφυρα με την, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, Σιγκαπούρης. Ορισμένοι από εσά, ο κ. Μάρτιν και λοιπά, έχουν επισκεφθεί την περιοχή αυτή και έχουν ε, δει τις ε, πρακτικές εκεί και ε, είναι πρόθυμοι να αξιολογήσουν τις αρχές που εφαρμόζονται εκεί, τόσο όσον αφορά την ε, κλιματική αλλαγή, της, ε, την απελευθέρωση του τομέα του εμπεριού κλπ. Ε, σε σχέση με το διεθνές δίκαιο και το πολυμερές σύστημα. Θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα πώς συνεργαστήκαμε στενά με το ILO ε, προκειμένου να ε, δημιουργήσουμε μια ασθενή ε, σχέση ένα, στη βάση ενός ειδικού προγράμματος ούτως ώστε να εφαρμόσουμε ένα κοινό πρόγραμμα ανάπτυξης στις χώρες Άζιαν και θα μπορούσα να σα δώσω πολλά άλλα παραδείγματα. Επιτρέψτε μου τώρα να μπω στο τρίτο μου σημείο να σας δείξω πώς οι δύο αυτές ε, συμφωνίε πραγματικά θα κάνουν τη διαφορά όσον αφορά όλου τους ενδιαφερόμενους και αξίζει να θυμηθούμε σαν μία από τις πλευρές που διαπραγματεύτηκαν τη συμφωνία. Τη συμφωνία αυτή είναι φιλόδοξη και ε, μακρόπνοη και θετική. Ε, πέρα από την απελευθέρωση και τα εμπερικά ωφέλη και αξίες, οι συμφωνίες συμπεριλαμβάνονται νέες καινοτόμες διατάξεις και συμπεριλαμβάνουν ε, μη δεσμολογικούς ε, φραγμούς. Θα μπορούσα να πω πολύ περισσότερα, αλλά θα σου δύο πολύ σύντομα παραδείγματα, ειδικά παραδείγματα. Η αλλάζει η Blue Solution υπέγραψε μια συμφωνία με τη Σιγκαπούρη, η πρώτη μεγάλη μεγάλης κλίμακας ε, συμφωνία για το σύστημα ε, ηλεκτρικής ε, τροφοδοσίας. Και υπάρχουν και πολύ επαρκείς κατευθυντήριες γραμμές τα νέα αυτοκίνητα ε, και τα νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα οποία θα ε, φτιαχτούν στη Σιγκαπούρη θα γίνονται άμεσα αποδεκτά Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω στον τομέα της ε, γεωργίας επίσης ε, υπάρχει ε, προβλέπεται η θέσπιση ενός συστήματος βάσει των ε, νέων συμφωνιών προκειμένου να διευκολυνθούν οι εισαγωγές ε, από γεωργικά προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Σιγκαπούρη. Η Ευρωπαίοι εξαγωγής ε, θα είναι πιο ανταγωνιστικοί από άλλους επιχειρηματίες που εξάγουν τα προϊόντα τους στην Σιγκαπούρη. Υπάρχουν πολύ περισσότερα παραδείγματα που θα μπορούσα να σας απεριθμίσω, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι ε, χρειάστηκε πολύς χρόνος να φτάσουμε σε αυτό το σημείο η κατάσταση τώρα είναι πολλά υποσχόμενη. Αναμένουμε λοιπόν την υποστήριξή σας για τις συμφωνίες αυτές προκειμένου να περάσουμε στην επιτυχή κύρωση και εφαρμογή εις όφελος ε, των εργαζόμενων τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των επιχειρήσεων ε, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην ε, Σιγκαπούρη. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα μας μένει μισή ώρα, δέκα άτομα ζήτησαν το λόγο και θα έχουμε επίση και μια παρέμβαση της ε, Επιτροπής ε, ε, καθώς και ερωταπαντήσεις. Ενάμιση λεπτό έχει ο κάθε ομιλητής, ο κύριος Κέλλη. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ και τους ομιλητές. Πιστεύω ότι τελευταία φορά που συζητήσαμε το θέμα αυτό ήταν πριν από 6-7 μήνες και ο κύριος Καμέλ είπε ότι ήταν ε, μια πολύ δυσάρεστη πρόταση ε, εκείνη την εποχή. Νομίζω ότι τώρα έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου να επικυρώσουμε αυτές τις ε, συμφωνίες. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν θέματα για τα οποία θα μπορούσαμε να παραπονεθούμε. Πραγματικά είναι ένα θαύμα αυτή οι συμφωνίες. Και υπάρχει μεγάλη δημιουργικότητα στην ε, Σιγκαπούρη. Πρόσφατα είχαμε και την επελέγη άλλωστε πρόσφατα για, να συναντηθούν εκεί οι ηγέτες Ηνωμένων Πολιτειών ε, και Βόρειας Κορέας. Ε, και θεωρώ ότι υπάρχει διακριτική μεταχείριση εδώ και της Σιγκαπούρης και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων γιατί έχουμε 10.000 ε, επιχειρήσεις που έχουν εκεί πέρα την έδρα τους και λόγω των επαφών που έχουν με ΙΠΑ, Κίνα και Ιαπωνία υποφέρουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οπότε πρέπει να ακυρωθεί αυτή η συμφωνία ε, τάχιστα και το υποστηρίζω 100%. Ε, ο κύριος Καμάλ, ευχαριστώ όπως ίσως ξέρετε πριν από πέντε χρόνια εγώ ήμουν εισηγητής, ο Ντέιβιντ ήταν σκιώδης εισηγητής και βεβαίως ε, μπορεί να διαφορούμε σε πολλά με τον Ντέιβιντ για το τι εστί η λογική κυβέρνηση. Συμφωνούμε ότι έχει καθυστερήσει αυτή η συμφωνία μαζί με τον κύριο Κέλλη άλλωστε. Και βεβαίω ε, όταν ε, συναντιούνται οι συγητέ, ε, συμφωνούμε όλοι και θέλουμε πραγματικά να προχωρήσει και είναι ντροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε απογοητεύσει την Σιγκαπούρη, αντιλαμβανόμαστε το πολιτικό ζήτημα και τους λόγους. Λοιπόν, θα σας κάνω κάποιες ερωτήσεις και αν έχετε χρόνο να απαντήσετε θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ. Το πρώτο είναι ότι είδαμε την παρουσίαση ναι, κάποιες ε, προβλέψεις ε, περί εμπορικών ροών και το τι θα συμβεί και στις ε, δύο πλευρές. Το 2003 ολοκληρώσετε την συμφωνία με τις ΗΠΑ και οπωσδήποτε τότε υπήρχαν κάποιες προβλέψεις. Αναρωτιέμαι λοιπόν εάν η πραγματικότητα ξεπέρασε τις προβλέψεις όσον αφορά την αύξηση των εμπορικών ροών ή όχι. Δεύτερον, προφανώς εμείς το ξανανοίξαμε το ζήτημα λόγω του μηχανισμού επίλυσης διαφορών. Τι σκέφτεστε λοιπόν με το CPTPP και το σχετικό κεφάλαιο εκεί και αν υπάρχει κάποια πιθανή σύγκρουση. Και βεβαίως έχω και ένα ευρύτερο ερώτημα για τον Αζίαν, αλλά νομίζω ότι είναι κάπως πρόωρο. Ευχαριστώ κύριε Στρεμόζα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, εξ ονόματος των φιλελευθέρων, θα ήθελα να πω ότι έχουμε καθυστερήσει για την έγκριση της συμφωνίας αυτής. Να σας υπενθυμίσω ότι ξεκινήσαμε το 2010, σταματήσαμε το 2013, ε, έπρεπε να ξαναδιαπραγματευτούμε, υπήρχαν διαφωνίες, έχουμε καθυστερήσει εν πάση περιπτώσει και θεωρώ ότι στην ομάδα μου υπάρχει κάποια απογοήτευση γιατί για την Ευρωπαϊκή Ένωση η συμφωνία αυτή είναι αμοιβαία επαφλής γιατί η Σιγκαπούρη είναι μια προχωρημένη οικονομία μια μικρή πόλη κράτος, ένας κόμβος για τις ευρωπαϊκές εταιρείες αλλά δεν παράγει γεωργικά προϊόντα ή κάτι άλλο που μπορεί να ανταγωνιστεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε λοιπόν μια ε, ανεπτυγμένη οικονομία που θέλει να αγοράσει προϊόντα από όλα τα κράτη-μέλη. Οπότε δεν καταλαβαίνω τους λόγους για τους οποίους ακόμα το συζητάμε. Και πραγματικά έχουμε κάτι το πολύ θετικό να πούμε στους πολίτες μας, να πούμε ότι κάνουμε κάτι χρήσιμο για αυτούς και για τις επιχειρήσεις μας. Και νομίζω ότι είναι και ένα καλό παράδειγμα για τις επόμενες ε, εμπορικές συμφωνίες, γιατί η Σιγκαπούρη έχει έναν ηγετικό ρόλο στις χώρες ε, του ΑΖΙΑΝ και πρέπει να δείξουμε στους πολίτες μας ότι είμαστε χρήσιμοι ως προς αυτό. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε για να μας δώσετε αυτές τις επιπρόσθετες πληροφορίες που θα μας χρησιμεύσουν στις χώρες μας και νομίζω ότι ε, θα υπάρχει μια ευρύτατη πλειοψηφία εντός του Κοινοβουλίου που θα εγκρίνει την συμφωνία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα αποτελέσματα αυτά της έκθεσης ε, είναι από το 2009 και βεβαίως ξεχνάμε ότι η Σιγκαπούρη βρίσκεται στην κορυφή όσον αφορά τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα κατά κεφαλή. Και πρέπει να δούμε τα θέματα τη κλιματική αλλαγή. Έχω δύο ερωτήσει. Λοιπόν, έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια πιο πρόσφατα αποτελέσματα για νούμερα για τα αποτελέσματα αυτή τη συμφωνία ε, επί του κλίματο. Και δεύτερον, σκοπεύετε να επαναλάβετε εδώ πέρα και την παράγραφο που υπάρχει στην ε, Συμφωνία της Ιαπωνίας για το κλίμα. Εάν όχι, γιατί όχι και αν ναι, τι μορφή θα έχει. Η Συμφωνία με τη Σιγκαπούρη λοιπόν έχει ε, ένα κεφάλαιο το οποίο λέει ότι θα παρακολουθείτε και από μια επιτροπή και από τους ενδιαφερόμενους και υπάρχει και μια ρήτρα αναθεώρησης ε, και βεβαίως θα υπάρξει και ένα πάνελ διατησίας από τρίτα μέρη, αλλά βεβαίως χωρίς κυρώσεις για τα πράγματα εκείνα τα οποία μας ενδιαφέρουν δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός καταναγκαστικός. Μετά, από τη μελέτη προκύπτει ότι ε, θα υπάρξει βλάβη για τις μικρές και μισές επιχειρήσεις, ε, ειδικά μετά όσα προβλέπονται για τους κανόνες ε, περί προέλευσης κατόπιν για την απόφαση του δικαστηρίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, βλέπουμε πώς αποσυνδέεται το κεφάλαιο για την προστασία των επενδύσεων από την εμπορική συμφωνία, ε, οπότε θα περιμένουμε την επόμενη απόφαση του δικαστηρίου για το κατά πόσο είναι συμβατό αυτό το σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Είναι διατεθειμένη η Κομισιόν να προσαρμόσει το χρονοδιάγραμμα για να περιμένουμε αυτήν την απόφαση. Και τέλος ε, δεν προβλέπεται το right to regulate, ε, ενώ υπήρχε στην ΙΣΕΤΑ. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί εξαφανίστηκε αυτός ο κανόνας. Ευχαριστώ. Τιτσιάνα Μπεγκίν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συνάδελφοι, εγώ όπως ε, ανέκαθεν έλεγα εδώ, πιστεύουμε στο εμπόριο όταν φέρνει ευημερία και ε, καλές συνθήκες ζωής, ε, όχι όταν χρησιμεύει ως ε, λεπίδα για να περικόπτει τα δικαιώματα των πολιτών. Και γι' αυτό και εγώ ίδια ενέκρινα την συμφωνία με την Ιαπωνία, αλλά και τώρα προτίθεμαι να εγκρίνω και αυτήν με την Σιγκαπούρη. Μιλώ για, για το ελεύθερο εμπόριο ε, είναι μικρή χώρα, αλλά από εκεί περνούν ε, πάρα πολλές ε, εξαγωγές και για τις υπόλοιπες χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ασίας. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει άνοιγμα ευκαιριών για αυτές τις αγορές. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και κάποιες ε, φαιές ζώνες ας πούμε συμπεριλαμβάνονται κανόνες για τη σώρευση του κανόνα προέλευσης που επιτρέπει να έρχεται από τη Σιγκαπούρη οποιοδήποτε προϊόν έχει εκεί παραχθεί και έχει την τελική του σφραγίδα από τη Σιγκαπούρη. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα σε προϊόντα ρουχισμού και σε τρόφιμα. Τώρα, μπορούμε να μιλήσουμε για εμπορική συμφωνία με τη Σιγκαπούρη, αλλά έχω πολλά προβλήματα με την ε, οδηγία, με τη συμφωνία ε, για την προστασία των επενδύσεων. Το ίδιο και η κυβέρνησή μου. Οι όμιλοι ε, μπορεί να έχουν ελευθερία για να ε, αντιπαρατεθούν στις κυβερνήσεις μας. Όπως και με την ε, ΣΕΤΑ και τη TTIP, δεν πιστεύω πως πρέπει να υπάρχουν τέτοιου είδη μηχανισμοί, διότι αυτή είναι επικίνδυνη για τη δημοκρατία και για τους πολίτες και εδώ είναι επίσης και άχρηστοι αυτοί οι μηχανισμοί αντίθετης των διαφορών. Ευχαριστώ. Μόιζερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστήσω τους συντάκτες της μελέτης που δείχνει οικονομετρικά ότι η συμφωνία θα είναι αμοιβαία υποφελής αυτό ήταν αναμενόμενο. Όμως για εμένα αυτό το οποίο δεν ποσοτικοποιείται είναι ακόμη πιο σημαντικό το ανάφερε ήδη ο Ντέιβιντ. Η Σιγκαπούρη είναι μια ασφαλής και προβλέψιμη χώρα για τις εταιρείες μας. Το πολιτικό μήνυμα που στέλνουμε σε έναν κόσμο που έχει προστατευτικές τάσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό αφορά την ταυτότητα και το πώς αυτό καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ε, ένας ε, παγκοσμίος ε, παίκτης και βέβαια στη Σιγκαπούρη έχουμε και μια υποχρέωση μετά από χρόνια βασανιστήριων για τους δικούς μας εσωτερικούς λόγους έχουμε υποβάλει την Σιγκαπούρη σε αυτή τη διαδικασία και θεωρώ ότι έχουμε υποχρέωση να συνάψουμε τη συμφωνία του στο Μοντρίνατον γι' αυτό ξαναρωτάω την Κομισιόν για το χρονοδιάγραμμα και αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος να μην ε, υπάρξει υπογραφή στις 19 Οκτωβρίου στο περιθώριο του ΑΣΕΜ. Για οποιονδήποτε λόγο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και τους εκπροσώπους ε, ε, της Σιγκαπούρης. Να σας ευχαριστήσω και για τη μεγάλη υπομονή που είχατε στη διάρκεια αυτών των μακρών διαπραγματεύσεων για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε. Νομίζω πως ήταν σκόπεμη η διαβούλευση ή μάλλον η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είναι σωστό να ε, χωριστούν οι δύο συμφωνίες αλλά βεβαίως ε, γι' αυτό το λόγο διέργεσε και τόσο πολύ περισσότερο αυτή η διαπραγμάτευση σε σχέση με την υπογραφή και την κύρωση των τριών θεμελιωδών συμβάσεων του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας που δεν, έχουν ακόμα, που δεν έχει ακόμα γίνει. Ελευθερία του συνεταιρίζεστε, η, αυτή που αναφέρεται στο εργατικό δυναμικό και τις διακρίσεις. Ε, και για τις τρεις συμβάσεις. Πρώτον, για ποιο λόγο η Σιγκαπούρη δεν τις έχει κυρώσει και ποιες είναι οι προοπτικές για την κύρωση αυτών. Δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με την ε, Συμφωνία Επενδύσεων που είναι μια μεγάλη ευκαιρία για, τις δυο, για τους δύο αλλά Εάν συνοδευτεί και από μια δυνατότητα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει να αναπτύξει όλες τις δυνατότητες. Από αυτή την προοπτική, ποια είναι η κατάσταση λοιπόν όσον αφορά την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων ε, στη Σιγκαπούρη των, ευρωπαϊκών ας πούμε, ε, πτυχίων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι μια στιγμή γλυκόπικρή γιατί όπως είπαν πολλοί συνάδελφοι ένα βασικό πρόβλημα της εμπορικής πολιτικής είναι ότι κρατάνε πολύ οι διαπραγματεύσεις και εδώ πέρα έχουμε πραγματικά ίσως την χειρότερη περίπτωση γιατί φταίμε εμείς. Και για τον λόγο αυτόν θεωρώ ότι αξίζει να το αναλογιστεί αυτό η Κομισιόν, το Συμβούλιο και οι συνάδελφοι εντός της εθούσης που δημιούργησαν αυτά τα προβλήματα. Γιατί ξεκινήσαμε με πολλές ελπίδες. Ξεκίνησε η διαπραγματεύση για τις υπηρεσίες και τα αγαθά το 2011. Εμείς θελήσαμε να προσθέσουμε το 2013 τις επενδύσεις. Ε, τα ολοκληρώσαμε όλα αυτά και ήθελε η Σιγκαπούρη να το υπογράψει αυτό, αυτή τη συμφωνία και μετά να συνεχίσουμε με την ε, συμφωνία περί επενδύσεων, αλλά αρνηθήκαμε τότε. Μετά το 2014 προσθέσαμε την ε, συμφωνία των επενδύσεων. Η Σιγκαπούρη είπε ναι, ναι, ωραία, να το υπογράψουμε. Μετά όμως το υποβάλαμε στο δικαστήριο, γιατί θεωρούσαμε ότι έπρεπε αυτή η συμφωνία να πάει στο δικαστήριο, ενώ ο Καναδάς δεν ήταν ζήτημα, μπορούσε να πάει στο Συμβούλιο και μετά εξέδωσε γνωμοδότηση το δικαστήριο, αλλά μετά θέλαμε να το ξαναανοίξουμε από την αρχή το κομμάτι των επενδύσεων. Και νομίζω πραγματικά ότι είναι ένα από τα χειρότερα παραδείγματα εμπορικής πολιτικής της Ένωσης και πρέπει να το ξαναδούμε αυτό και να πούμε ότι δεν θα ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Πρέπει λοιπόν να μην έχουμε πια άλλα εμπόδια. Το μόνο το οποίο άκουσα από τους συναδέλφους είναι ότι κάποιοι συνάδελφοι ανησυχούν για τις ε, συμβάσεις του ΑΕΛΟ. Θα ήθελα να μάθω αν υπάρχουν πραγματικές ανησυχίες, πείτε τα τώρα, αλλιώς μην ξαναμιλήσετε. Ή αν είναι απλά κάτι το οποίο θέλετε να κάνετε τυπικά. Σας παρακαλώ δηλαδή, όχι άλλα εμπόδια. Καρολίν, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, παρουσίαση και την επισκέψή σας κύριε Γκο η απόφαση του δικαστηρίου χρειάστηκε λίγο καιρό, αλλά ε, νομίζω ήταν χρήσιμο το να ξέρουμε τι μπορούμε να αποφασίσουμε. Όπως είπαμε, η Σιγκαπούρη είναι κόμβος στην Ανατολική Ασία, έχει υψηλές προδιαγραφές, γι' αυτό ακριβώς ε, το ερώτημα είναι ε, γιατί δεν έχουν ακόμα κυρωθεί οι συμβάσεις του Άιλο ποιοι είναι οι λόγοι. Μιλάμε για τα ελάχιστα τα οποία δεν θα έπρεπε να αποτελούν πρόβλημα για την ε, Σιγκαπούρη και κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω όσον αφορά το θέμα της αηφορίας και αν δεν υπάρχουν κυρώσεις, ποιοι μηχανισμοί υπάρχουν τότε όταν έχουμε παραβιάσεις ε, των διατάξεων για το περιβάλλον, ποιες δυνατότητες υπάρχουν, γιατί εμείς θέλουμε συμφωνίες δίκαιες που θα βασίζονται σε κανόνες και θεωρούμε ότι ένα κεφάλαιο για την εφορία μπορεί να είναι ισχυρό μόνο αν υπάρχουν και κυρώσεις. Σας ευχαριστώ, Βίνκλερ. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες αυτές. Ε, δύο σημεία θα ήθελα να αναφέρω. Το παγκόσμιο πλαίσιο και την ρεαλιστική προσέγγιση που απαιτείται. Βεβαίως, θα ήθελα εδώ πέρα να επενέσω και τον David Μάρτιν και η παγκόσμια σημασία αυτής της συμφωνίας έχει πολλές διαστάσεις γιατί έχουμε την πρώτη συμφωνία με μέλος του ΑΖΙΑΝ αλλά έχουμε και το παγκόσμιο πλαίσιο ε, κάποιες χώρες ε, φτιάχνουν είχε εμείς θέλουμε να φτιάξουμε γέφυρες ε, μίλησαν για τη συνδεσιμότητα οι συναδελφοί από την Σιγκαπούρη. Πράγματι αυτό έχει μεγάλη σημασία τον 21ο αιώνα και να επαναβεβαιώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανοιχτή για τις επιχειρήσεις. Και έρχομαι άρα στο δεύτερο σημείο, την ρεαλιστική προσέγγιση που απαιτείται. Και εδώ πέρα έχουμε τον Κριστόφ Φιέλνερ που λέει πως θα πρέπει ακριβώς να θέλουμε τις υπογραφές και όχι μια προσωρινή εφαρμογή και να μην έχουμε κανένα εμπόδιο που θα μπορούσε να σταθεί ε, μπροστά στην, ε, και να εμποδίσει την προσωρινή εφαρμογή. Ακριβώς για να ανακτήσουμε την αξιοπιστία μας απέναντι στους παγκόσμιους εταίρους μας. Και το ερώτημά μου είναι πως η Κομισιόν έχει γίνει ήδη, είναι πάρα πολύ απλό, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, εάν μπορείτε να το μοιραστείτε μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπαν ήδη οι συνάδελφοι, η ιστορία της εμπορικής συμφωνίας και της συμφωνίας για την προστασία των επενδύσεων με τη Σιγκαπούρη είναι πολύ μακρά, υπερβολικά μακρά ίσως και είναι το πρώτο που θα έπρεπε να πούμε στους εταίρους μας στη Σιγκαπούρη. Σας ευχαριστούμε για την τεράστια υπομονή σας, την καλή σας προαίρεση και την επικοδομητική σας προσέγγιση. Και πιστεύω ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για την Ευρωπαϊκή Ένωση να μείνει πιστή στους εταίρους της, δηλαδή να ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία. Βεβαίως, μετά από όλο αυτό το καιρό, οι συμφωνίες αυτές παραμένουν όπως είπα, στρατηγικά σημαντικές, οικονομικά ισορροπημένες και διανοίγουν νέες ευκαιρίες και για τις δύο πλευρές. Και νομίζω ότι αυτό είναι παραπάνω από αρκετό. Και είναι αλήθεια ότι μεταξύ πολλά πράγματα έχουν αλλάξει στο παγκόσμιο εμπόριο και στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάπως ε, καθιστούν ε, δύσκολο να αξιολογήσουμε συμφωνίες που έχουν διαπραγματευτεί πριν από μερικά χρόνια, αλλά με βελτιώσεις που θα γίνουν ε, στις συμφωνίες, τελευταία φάση διαπραγμάτευση, μπορούμε να πούμε, όπως ε, είπε και ο συγητής κ. Μάρτιν, ότι σε πολλούς ε, τομείς έχουμε πιο προοδευτικές λύσεις τώρα από αυτές που έχουμε για την ΣΕΤΑ. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένας λόγος να αναβληθεί η απόφαση αυτού του Κοινοβουλίου ε, λαμβάνοντας ε, υπόψη ότι αυτό δεν είναι το τέλος όλης της ιστορίας και οι συμφωνίες ε, μπορούν και πρέπει να βελτιωθούν και μελλοντικά και το να μιλάμε για βελτιώσεις στους φίλους από την Σιγκαπούρη συνεπάγεται και την κύρωση των διατάξεων των, ε, του ΑΕΛΟ. Ε, ε, μόνο θα, θα ήθελα να πω, να επισημάνω στον κύριο Φέλμερ ότι το γεγονός ότι θέλει να γνωρίζει επακριβώς την εμβέλεια που έχουν αυτές οι συμβάσεις του ΑΕΛΟ, που βρίσκονται στον πυρήνα των εργασιακών συμβάσεων το να ε, νομίζω ότι ε, είναι αναγκαίο το αίτημα να τις ε, διεκδικήσουμε. Ευχαριστούμε και τώρα θα ήθελα να καλέσω τον Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου να, την κυρία Μαρία Θράτη, να σχολιάσει από την δική της πλευρά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολλές ε, παρατηρήσεις έγιναν σε σχέση με τον ε, μεγάλο μακρύ χρόνο αυτών των διαπραγματεύσεων και την υπομονή που έδειξαν όλοι οι ενεχόμενοι στην διαπραγματευτική διαδικασία που δίερκησε υπερβολικά πολύ. Και η Επιτροπή δεν μπορεί να συμφωνήσει με όλα αυτά και θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τη Σιγκαπούρη για το ζήλο που επέδειξε και την υπομονή της. Ε, ε, εγώ ήμουν ε, επιφορτισμένη για τον διαχωρισμό της συμφωνίας σε δύο μέρη. Αυτό ακλά στην ανάγκη μιας νέας αρχιτεκτονικής εν ώψη και εν ώψη του ότι έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό είναι μια επιτυχία. Ε, οι συμφωνίες αυτές ε, σήμερα είναι πιο σημαντικές ακόμα από ό,τι υπήρξαν, ήταν όταν ε, πρώτη φορά συνέφθησαν πριν από πέντε χρόνια. Δυστυχώς όμως ο κόσμος, το παγκόσμιο σκηνικό άλλαξε με έναν τρόπο που είναι πιο σημαντικό για μας να έχουμε έναν εταίρο όπως είναι η Σιγκαπούρη ε, για ένα δίκαιο και θεμητό εμπόριο, θεμητές και δίκαιες εμπορικές συναλλαγές στην περιοχή. Γιατί η Σιγκαπούρη παίζει εδώ ένα καθοριστικό ρόλο σε πολυμερές επίπεδο. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να φωτίσω είναι το γεγονός ότι με τις δύο αυτές συμφωνίες έχουμε μια ότι μπορούμε να μεταφέρουμε στην περιοχή αυτή τα πρότυπά μας όσο αφορά το εμπόριο και τα πρότυπά μας όσον αφορά την προστασία των επενδύσεων όπου ο ε, συγητής ε, ε, είπε ότι υπάρχει το υπόδειγμα της ΣΕΤΑ, περιλαμβάνοντας στοιχεία διαφάνειας και δικαίου όσον αφορά την προστασία των επενδύσεων, εις όφελος των επενδυτών μας, αλλά με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων της άλλης πλευράς. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε μια εποχή όπου ε, προδιαγραφές παραβιάζονται από άλλους. Έχει ήδη αναφερθεί η CPTPP και συνεχιζόμενες ε, διαπραγματεύσεις είναι σημαντικό η Ευρώπη να έχει τις δικές της προδιαγραφές στην περιοχή αυτή, η οποία είναι ε, ιδιαίτερα σημαντική κατά την άποψή μας και με την, όσον αφορά το εμπόριο με τη Σιγκαπούρη και με την ε, Συμφωνία για την Προστασία Επενδύσεων ε, εδραιώνουμε την παρουσία μας στην περιοχή και αυξάνουμε την αξιοπιστία μας και θεωρούμε ότι είναι μια πρώτη συμφω... διμερή συμφωνία επενδύσεων και εμπορίου με μια χώρα στην περιοχή αυτή, πράγμα που είναι τεράστια σημασία όσον αφορά την αξία της Σιγκαπούρης ως εταίρου ένα τρίτο του εμπορίου και ένα μεγάλο μέρος επενδύσεων αφορούν τη Σιγκαπούρη στην περιοχή αυτή. Παρ' όλα αυτά, ο στόχος ε, βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να συνάψει συμφωνίες και να κάνει επενδύσεις ε, σε ολόκληρη την ε, περιοχή αυτή, όχι μόνο στη Σιγκαπούρη. πολλοί αμελητές επεσήμεναν κάποια προβλήματα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και είμαι πεπισμένη ότι και η Συγκαπούρη έχει δεσμευτεί να κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να αποφευθούν ε, ε, ενδεχόμενα προβλήματα, να μην σκαλώσουν τα πράγματα. Ε, εμείς θέλουμε να επισπεύσουμε τις ε, προσπάθειες στο επίπεδο του Συμβουλίου και της Συγκαπούρης. Υπάρχουν προθεσμίες για τις χώρες μέλη να σχολιάσουν για τα σχέδια των συμφωνιών το καλοκαίρι. Στην αρχή Οκτωβρίου το Συμβούλιο θα εγκρίνει τις αποφάσεις και θέλουμε να έχουμε την υπογραφή της συμφωνίας στη συνάντηση κορυφής ΕΖΙΑΝ στον, στα μέσα Οκτωβρίου και στη συνέχεια θα αποσταλεί στο Κοινοβούλιο για να δώσει την δική του συγκατάθεση. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Ε, ε, ε, εργαζόμαστε με μεγάλη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, ούτως ώστε να μπορέσει να υπογραφεί συμφωνία τον Οκτώβριο. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Κύριε Ρουσό, θέλετε να σχολιάσετε. Κυρία Ρουσό, συγγνώμη, θέλετε να σχολιάσετε. Νομίζω ότι εναπόκειται στην ε, Κομισιό να απαντήσει. Κύριος... Γκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την στήριξη και την προσήλωση που επιδείξατε για να προχωρήσει η συμφωνία. Πράγματι αναγνωρίζω και εγώ τα ερωτήματα τα οποία θα προσπαθήσω να απαντήσω ειδικά για τα ζητήματα του Διεθνούς Γραφείου Εργασία. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε πιο αναλυτικά για να σας εξηγήσω, όχι για ζήτημα ψήφων, αλλά να σας εξηγήσω τα ζητήματα αρχής, ε, γιατί είναι σημαντικό το θέμα των εργασιακών δικαιωμάτων, όχι μόνο για εσάς, όχι μόνο για τη Σιγκαπούρη, αλλά και για εσάς. Ε, γιατί το ανέφερε και ένας συνάδελφος, να μην είναι κάτι το τυπικό. Λοιπόν, για όλα τα άλλα ζητήματα να αναφερθώ. Ο κύριος Καμάλ π.χ. αναφέρθηκε στο ε, πώς ε, μεταφράστηκαν στην πράξη οι προηγούμενες συμφωνίε ελευθερίου εμπορίου, παραδείγματο χάρη με τις ΗΠΑ. Ουσιαστικά στα χρόνια ε, ισχύω αυτή τη συμφωνία έχουν διπλασιαστεί οι εμπορικέ ε, ροές και οι επενδύσει επίσης έχουν πολλαπλασιαστεί και επίσης υπάρχει και το ζήτημα καθορισμού των κανόνων και βεβαίως τώρα έχουμε και την συμφωνία TPP Οπότε βεβαίως δεν ξέρουμε τι μπορούμε να αποδώσουμε μόνο στη Συμφωνία Ελευθερού Εμπορίου, αλλά θα έλεγα ότι αποτέλεσε αφετηρία για πάρα πολλές ε, θετικές εξελίξεις ε, και βεβαίω και βασικό είναι το ότι έχουμε μια πλατφόρμα συνεργασίας και επίλυσης διαφορών. Μετά υπάρχει το ζήτημα που ετέθη για τον μηχανισμό επίλυσης ε, διαφορών. Πρώτα απ' όλα από την σκοπιά της Σιγκαπούρης εμείς δεν βλέπουμε κάτι το αντιφατικό να προκύπτει από τις υποχρεώσεις μας για τα συστήματα αυτά προστασίας των επιμήσεων. Βεβαίως προτιμούμε να έχουμε ένα σύστημα, τελικά καταλήξαμε στο ICS χωρίς ε, καμία αμφιβολία, δεν είχαμε καμία φιλοσοφική ε, αντίρρηση, οπότε τώρα έχουμε το ICS, αλλά Τελικά, εάν ο κόσμος μπορεί να προχωρήσει σε ένα πολυμερές τέτοιο σύστημα, αυτό θα αποτελούσε έναν μεγάλο βαθμό διαφάνειας. Ε, υπήρξε όμως ένα σχόλιο για το πώς, αν ε, υπάρχει όντως ανάγκη ε, για ένα τέτοιο σύστημα μεταξύ ανεπτυγμένων οικονομιών και η απάντησή μου βεβαίως ε, είναι δίτη. Ρωτήστε τις εταιρείες, ε, τις ευρωπαϊκές εταιρείες όταν έρχονται στην Σιγκαπούρη και στην περιοχή γενικότερα εάν θέλουν έναν τέτοιο μηχανισμό. Δεν αγγινάνε να είναι ISDS, μπορεί να είναι ICS ή κάτι άλλο. Θα σας πούν νομίζω ότι όσο είναι στην Σιγκαπούρη δεν έχει υπάρξει καμία ε, αμφισβήτηση. Και ισχύει και το αντίστροφο βεβαίως με τις εταιρείε μας στην Ευρώπη, αλλά στην υπόλοιπη περιοχή ε, καλύτερα να σας τα πούν οι ίδιες οι εταιρείε, αλλά νομίζω ότι θα σας πούν ότι έχει μεγάλη αξία για τις εταιρείε ε, και αντιστρόφως για τις επενδύσεις της Σιγκαπούρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν το χρειαζόμαστε. Η απάντηση είναι όχι, γιατί ποτέ δεν έχουμε βρει κάποιον λόγο διαμάχης, αλλά επειδή η ανησυχία σας μπορεί να προέρχεται από το εάν θέλετε μεγάλες εταιρείε να λαμβάνουν ορισμένες λειτουργίες. Ρωτήστε τις ευρωπαϊκές εταιρείε ε, και τους δικούς σας, το προσωπικό σας που έχει κάποια σχέση με την αγορά της Σιγκαπούρης, εάν υπάρχει κάποια εταιρεία της Σιγκαπούρης αρκετά μεγάλη για να παίξει τέτοιο ρόλο στην ευρωπαϊκή αγορά. Μιλάμε για μια χώρα 3,5 ε, εκατομμυρίων έχουμε κάποιες εταιρείε όπως η Singapore Airlines ε, οπότε σας ε, διαβεβαιώ ότι δεν είμαστε κάποιο είδους απειλή και σκεφτείτε το αυτό. Και τώρα νομίζω μπορούμε να περάσουμε στα θέματα του ILO. Να δηλώσω ξεκάθαρα πως είμαστε προσιλωμένοι σε υψηλές ε, προδιαγραφές όσον αφορά τα εργασιακά. Δεν είναι λόγια μόνο αυτά και ε, Γενικός Διευθυντής του οργανισμού νομίζω μπορεί να βεβαιώσει την πρόοδο που έχουμε σημειώσει. Είπατε πως ε, οι συμβάσεις αυτές είναι κάτι το βασικό και πράγματι σε πολλές περιπτώσεις το έχουμε ξεπεράσει. Αλλά το ερώτημά σας είναι γιατί δεν έχουμε κυρώσει κάποιες. Ε, υπάρχουν δύο παράγοντες ε, που μας κάνουν να είμαστε κάπως επιφυλακτικοί. Ο πρώτος παράγων είναι εξής, ότι ε, κοιτάμε τα αποτελέσματα πρώτα απ' όλα και από οποιοδήποτε καθεστώς, οποιαδήποτε σύμβαση, αν οδηγεί στα θετικά αυτά αποτελέσματα για τους εργαζόμενους. Ποια είναι αυτά τα αποτελέσματα λοιπόν. Μιλάμε για το ποσοστό απασχόλησης, ε, το εισόδημα ανακεφαλή και όπως σας είπα με λιγότερα από 4 εκατομμύρια πολίτες είναι υπαρξιακό ζήτημα για μας να φροντίσουμε να μην υπάρχουν διαμάχες εργασιακές, να έχουμε ακριβώς μια τριμερή συνεννόηση εργαζομένων, κράτους και συνδικάτων. Και αυτή είναι η απάντηση ακριβώς για το ότι δεν υπάρχουν αυτές οι παραβιάσεις που ε, πιθανώς Γιατί ε, προσπαθούμε να μην υπάρχει κάποια διαμάχη γιατί ακριβώς αναζητούμε κάποια πλατφόρμα η οποία θα είναι είτε κρατική είτε οτιδήποτε άλλο. Αλλά στο σύστημα της Συγκαπούρης, το σύστημα της Συγκαπούρης είναι τριμερές. Έχουμε λοιπόν το κράτος και τα συνδικάτα και τα συνδικάτα είναι ισχυρά. Πρέπει να δω τον, τον ακριβή αριθμό, αλλά ε, είναι διψήφιος σίγουρα ε, και έχουν ε, αρκετά μεγάλη επιρροή. Ελάτε στην Σιγκαπούρη ε, και ευχαρίστω ε, να σας τα δείξουμε. Γιατί ακριβώς δεν εμπίπτει στον δικό σας τον ορισμό. Γιατί τα συνδικάτα είναι ήδη μέρος του μηχανισμού διαιτησίας και προσφυγής. Λοιπόν, για να επανέλθω. Η Σιγκαπούρη έχουμε μια φήμη να προστατεύσουμε και οτιδήποτε υπογράφουμε το εφαρμόζουμε 100%. Αν λοιπόν είμαστε αβέβαιοι για κάτι το συζητάμε και το εξετάζουμε προσεκτικά. Όταν μιλάμε λοιπόν για τις ε, συγκεκριμένες ε, συμβάσεις. Γνωρίζετε ότι οι συμβάσεις είναι μακροσκελή κείμενα με πολλές υποχρεώσεις ε, και μεγάλο βαθμό λεπτομέρειας. Και βρίσκομαι εδώ να σας πω το εξής. Σήμερα νωρίτερα υπήρχε και μία συνεδρίαση με την ε, κυρία Βαργκάς ε, του ILO, την Διευθύντρια, και είπαν οι ίδιοι ότι ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι οπωσδήποτε έχουν υπογράψει όλες τις συμβάσεις, πόσο σίγουροι είστε ότι όλα αυτά, οποιαδήποτε λεπτομέρεια των συμβάσεων εφαρμόζεται πλήρως. Και ήταν ένα ρητορικό ερώτημα. Για την Σιγκαπούρη λοιπόν, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να ελεγχθούμε σε οτιδήποτε έχουμε υπογράψει. Γιατί λοιπόν δεν υπογράφουμε και τις υπόλοιπες δύο-τρεις ε, συμβάσεις. Πρώτα απ' όλα μία από τις συμβάσεις ε, που λέτε ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να εισαχθεί μία νομοθεσία μη διακριτικής μεταχείρισης. Σήμερα έχουμε ένα καθεστώς που αποθαρρύνει τη διακριτική μεταχείριση ε, διάφορα συστήματα και αυτό γίνεται και ελέγχεται όχι μόνο από κρατικές υπηρεσίες και πάλι τα συνδικάτα συμμετέχουν σε αυτό. Το κάνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Γιατί λοιπόν να μην το επισημοποιήσουμε. Ε, γιατί σε μια πολυφιλετική, πολυεθνική κοινωνία, κάτι το οποίο πρέπει να αντιλαμβάνεστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ένα σύστημα σαν το δικό μας, δεν θέλουμε να πούμε ότι τώρα όταν κάποιος ζητάει μία θέση ε, χρειάζομαι κάποιον ο οποίος μιλάει την γλώσσα την ε, κινέζικη ή την ε, ταμίλ γιατί συχνά αυτό προβλέπει ο νόμος τον οποίο θέλετε. Δεν θέλουμε λοιπόν να έχουμε τέτοια νομοθεσία. Αν δείτε όμως τον σκοπό της σύμβασης στην ουσία τον εκπληρώνουμε. Η απάντηση είναι ναι, αλλά εμείς δεν θέλουμε να ε, χάσουμε αυτήν την ε, ευελιξία. Να σας δώσω άλλο ένα παράδειγμα και θα τελειώσω. Έχουμε ε, ακριβώ κάτι άλλο το οποίο απαγορεύει τα προγράμματα εργασία τη φυλακή. Οι φυλακές μας είναι ανοιχτές σε ΜΚΟ που έχουν έρθει και μας έχουν επενέσει για το πρόγραμμα αυτό το πρόγραμμα, το, ποσοστό επίσης επανένταξης ε, ή αν θέλετε υποτροπής μετά είναι από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο στον κόσμο. Αυτά τα λένε διάφορες ΜΚΟ που έχουν έρθει και τα έχουν δει. Αυτό σημαίνει όμως ότι πρέπει να έχουμε προγράμματα εργασίας και κατάρτισης στις φυλακές. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι ε, το πρόγραμμα αυτό παραβιάζει τις ε, συμβάσεις Οπότε, εάν υπογράψουμε την σύμβαση, θα πρέπει να σταματήσουν κάποια αυτά. Είναι ένα μέρο μια αλυσίδα και δεν αφορά μόνο τι ε, φυλακέ, αφορά και την απασχόληση εκτό των φυλακών ή με το ότι οι πρώην κρατούμενοι πάνε στις φυλακές και μιλάνε στους νυν κρατούμενους ε, κτλ. Υπάρχουν νομίζω πολλές ε, χώρες που θα έκαναν κάτι τέτοιο και δεν θα ακούγαν τέτοια κριτική. Λοιπόν, επειδή η χώρα μας έχει επιλέξει να είναι πολύ τυπική στους κανόνες ε, σε οτιδήποτε υπογράφουμε, ε, τώρα ε, τιμωρούμαστε γι' αυτό. Δηλαδή το θέμα είναι και το τι γίνεται στην πραγματικότητα. Μην ακούτε εμένα. Λάτε να δείτε το τι γίνεται στην πράξη και κρίνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. David, μπορείς να κλείσεις. Ναι, θα είμαι σύντομος. Πρώτον, είναι νομίζω ευρία η στήριξη της Επιτροπής για αυτή τη συμφωνία και ε, στηρίζω τα όσα είπα και η Κομισιόν ότι είναι πιο σημαντική από ό,τι ήταν πριν πέντε χρόνια όταν αρχικά χρειάστηκε να παγώσουμε τη συμφωνία. Και αυτό λόγω της παγκόσμιας κατάστασης που συζητήσαμε και όλοι τη γνωρίζουμε. Επειδή έχω επισκεφθεί μια-δύο φορές στη Σιγκαπούρη και μελέτησα κάποια από τα θέματα για τα οποία μόλις μιλήσατε κύριε Γκουάου, ε, ε, συμφωνώ ότι κάποιες φορές η Σιγκαπούρη τιμωρείται επειδή είναι υπέρ του κράτους δικαίου. Πολύ υπέρ. Και φροντίζει πάντα να εφαρμόζονται όλα πλήρως. Αν δείτε κάποιους ε, γείτονες που χαροπά υπέγραψαν τις συμβάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, δεν τις εφαρμόζουν. Η Σιγκαπούρη λάμπει, είναι αστέρι σε σχέση με τους γείτονές της. Θα σας δώσω και περισσότερες πληροφορίες για γιατί δεν έχουν υπογραφεί οι τρεις συμβάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την υπογραφή αυτών των ε, συμβάσεων. Πρέπει να καταλάβουμε γιατί δεν υπογράφηκαν. Τώρα, επίσης σωστά θέσατε το θέμα του περιβάλλοντος. Και αν δείτε το κείμενο, το τμήμα για το περιβάλλον είναι αρκετά εθαρρυντικό βέβαια, θα πρέπει να εφαρμοστούν και τα όσα λέει. Πάντως το ίδιο το κείμενο είναι καλό. Εν γέννη, η Σιγκαπούρη είναι μία από τις χώρες που έχει δεσμευθεί σε 36% μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα μέχρι το 2030. Και εκεί υπάρχουν δύο συγκεκριμένα τμήματα για τις επενδύσεις και το εμπόριο όσον αφορά την ανανεώσιμη ενέργεια. Οπότε... Ε, αυτό το θέμα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν ε, με το, μέσο του εμπορίου και υπάρχει και ένα γενικότερο τμήμα για το πώς ε, περίπου 10 παράγραφοι για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Σιγκαπούρη μπορούν να συνεργαστούν ώστε να ε, γίνουν προσπάθειες πάντα σε σχέση με το εμπόριο. Αναγνώριση των επαγγελματικών δεξιοτήτων είναι επίσης στο τμήμα 816, αυτό που ρωτήσατε. Υπάρχουν κάποιες τοπικές εξαιρέσεις, αλλά εν γέννη ε, έχουμε σκεφτεί και έχουμε τονίσει την αμοιβαία αναγνώριση. Η ανησυχία μας για τις επενδύσεις δεν αφορούν το πώς θα λειτουργήσει το κεφάλαιο για τις επενδύσεις. Μια εταιρεία που λειτουργεί στη Σιγκαπούρη θα μπορεί να κάνει ενέργειες και η Σιγκαπούρη δεν είχε ποτέ μια διαμάχη περί επενδύσεων μέχρι στιγμής, οπότε η πιθανότητα να προκαλέσει διαφορές αυτή η συμφωνία είναι μάλλον ισχνή. Νομίζω πάντως ακούσατε ότι η διπλοψηφία του Κοινοβουλίου φαίνεται ε, να αισθάνεται ένοχη για το ότι καθυστέρησε αυτή η συμφωνία και θέλουμε να ολοκληρώσουμε την έγκριση. Ε, μέχρι που να υπογραφεί τον Οκτώβριο έχουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να περάσει γρήγορα από το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. So, dear colleagues, the last item on our agenda is the implementation report on the trade Τελευταίο σημείο στην ημερησία μας διάταξη είναι η εκθέση εφαρμογή σχετικά με τον εμπορικό πυλώνα της Συμφωνίας σύνθεσης με την Κεντρική Αμερική και θα έχουμε ακριβώς 20 λεπτά. Παρακαλώ, ησυχία. Yeah. Yeah. So, exactly 20 minutes. You know this... 20 λεπτά γιατί γνωρίζετε την κατάσταση με τους διερμηνείς. Ε, δεν δίνουν ε, υπέρβαση ωραρίου ε, λόγω της διαμαρτυρίας τους που συνεχίζεται. Ευχαριστώ Πρόεδρε, λέει ο κ. Μπέγκη, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Θα ξέρετε ότι υπογράφηκε συμφωνία σύνδεση με την Κεντρική Αμερική το Σεπτέμβριο, το Δεκέμβριο του 2012 εδώ. Υπογράφηκε, ήταν η πρώτη περιφέρεια που έφτιαξε τέτοια συμφωνία και πρόκειται για τρεις πυλώνες πολιτικό διάλογο, συνεργασία και εμπόριο. Βεβαίως η εκθέση εφαρμογής εστιάζεται στο πυλώνα του εμπορίου. Και υπάρχουν και κάποια θέματα που αφορούν το εμπόριο ε, στους άλλους δύο πυλώνες. Ο πυλώνας του εμπορίου έχει, έχει εφαρμοστεί εδώ και πέντε χρόνια από τον Αύγουστο του 18 από τους εταίρους μας της Κεντρικής Αμερικής. Θέλω μόνο να πω ότι προετοιμάζοντας αυτή την ανταλλαγή απόψεων σήμερα είχαμε μία επαφή με τους ε, εκπροσώπους της Λατινικής Αμερικής με τη συμμετοχή της DG ε, ε, Trade και τον εκπρόσωπο των πρέσβη της Κωνσταντίνα που έχει την κυλιόμενη Προεδρία για τους τελευταίους έξι μήνες. Η, έκθεση, ε, η έγκριση της έκθεσης προβλέπεται για το Δεκέμβριο. Λοιπόν, καταρχάς ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτής της συμφωνίας σύνδεσης για τις δικές μας εμπορικές σχέσεις. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Κομισιόν από τον Νοέμβριο του 2017 για την εφαρμογή ε, της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου θεωρήθηκε πως έχει σταθεροποιητικό ε, εφέ για το διμερές εμπόριο Ένωσης Κεντρικής Αμερικής ήταν σταθερό, δεν αυξήθηκε οι συναλλαγές, αλλά παρέμειναν σταθερές παρά τις δυσμενείς διεθνείς συνθήκες. Είχαμε κάποιες ενδιαφέρουσες στατιστικές από την Κομισιόν που μας λένε ότι εξακολουθεί να υπάρχει κάποιο περιθώριο ελιγμού. Για παράδειγμα, για τη ζάχαρη οι ποσοστώσεις ε, απορροφήθηκαν τελείων, ενώ κάποια άλλα προϊόντα δεν το χρησιμοποίησαμε πλήρως και από τις δύο πλευρές. Έχουμε να κάνουμε επίση με τις εξηγήσει στην έκθεση αυτή, για ποιο λόγο ας πούμε έγιναν όλα αυτά. Όταν δούμε τα κύρια προϊόντα που εξάγονται από την Κεντρική Αμερική προς την Ένωση, έχουμε μεγάλη συγκέντρωση στον τομέα των τροφίμων, ας πούμε καφές, μπανάνες, ε, ε, ε τόνος κονσέρβα και εξάγουμε και προϊόντα με περισσότερη προστιθέμενη αξία όπως ε, προσθετικές ε, συσκευές, ιατρικές συσκευές ε, και για βιολογικά προϊόντα που έχουν την πιστοποίηση Fair Trade. Οι βασικές εξαγωγές από την Ένωση είναι φάρμακα, αυτοκίνητα, ανοσοποιητικά προϊόντα, ουίσκι, κοσμήματα και διάφορα άλλα. On the FDI flows. Αν δούμε τις ροές, έχουν αυξηθεί και από τις δύο πλευρές. Αυτή τη στιγμή υπολογίζονται σε 26 δις ευρώ για την Ένωση και 11 δις ευρώ για την Κεντρική Αμερική. Για την εφαρμογή Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε λάβει από τις ομάδες παρακολούθησης, το γενικό επίπεδο δεσμεύσεων από, υποχρεώσεων από την, από την Κεντρική Αμερική είναι κατοπιτικό. Πολλά ζητήματα SPS ε, έχουν επιληθεί Επίσης, το ίδιο όσον αφορά τις ε, διαδικασίες για τη συνεργασία έχουν βελτιωθεί ώστε να είναι πιο προβλέψιμη η κατάσταση για τους Ευρωπαίους επιχειρηματίες. Υπάρχουν κάποια ερωτηματικά για τη φορολόγηση του αλκοόλ καθώς και για τις παραβιάσεις ε, των... της περί ανταγωνισμού στην Κωνσταντίνα και στην Νικαράγουα. Επίσης, θέματα εργατικά Ονδούρα, Γουατεμάλα, Ελσαλβαδόρ Ίσως να έχουμε περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σήμερα ε, ή την επόμενη φορά που θα υποβάλλει η Κομισιόν έκθεσή της. Μεγάλη σημασία είναι βέβαια το γεγονός ότι οι διεθνείς προδιαγραφές για το περιβάλλον και την απασχόληση να εφαρμόζονται πλήρως. Να τονίσω ένα κρίσιμο σημείο που είναι λυπηρό και πάλι, είναι το ότι θα ήθελα να καλέσω τα ευρωπαϊκά κράτη να κυρώσουν αυτή τη συμφωνία ώστε να μπει σε εφαρμογή πλήρως η συμφωνία. Λείπουν το Βέλγιο, η Αυστρία, η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο που δεν έχουν ολοκληρώσει την εσωτερική διαδικασία τους. Ενώ από την άλλη πλευρά η Κεντρική Αμερική έχει κάνει τη δουλειά της για να διευκολύνει την προσχώρηση της Κροατίας σε αυτή τη συμφωνία. Και πάλι λοιπόν πρέπει να επιμείνουμε προς τα κράτη-μέλη και τα εθνικά τους κοινοβούλια να κυρώσουν τη συμφωνία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ναι, θα το πω σήμερα και όλα, το, είπα και όλα στον Υπουργό της Αυστρίας σήμερα, αλλά πρέπει να πιέσουμε. Χωρίς μικρόφωνο η ομιλήτρια. Άμεση perdón να τα ξαναπώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και σας ε, κύριε Συγητή, για τη λεπτομερή εισήγηση που μας κάνατε σε σχέση με τη Συμφωνία για την Κεντρική Αμερική και την εφαρμογή της. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω με τα τελευταία σας λόγια, να συμφωνήσω με αυτά που είπατε στην ε, Αυστριακή Προεδρία σήμερα το πρωί, την ανάγκη κύρωση της ε, συμφωνίας και του του πολιτικού διαλόγου συνεργασίας από πλευρά των κρατών μελών, γιατί μάλιστα οι περιστάσεις που επικρατούν σε κάποιες χώρες της Κεντρικής Αμερικής έχουν καταστήσει αυτή τη συμφωνία πιο απαραίτητη από ποτέ. Η συμφωνία αυτή βασίζεται σε τρεις πυλώνες και είναι θεμελιώδες η πολιτικός διάλογος συνεργασίας να ενισχύσει την, ε, τον εμπορικό πυλώνα ώστε να βοηθήσουμε στην βιώσιμη ανάπτυξη. Θα ήθελα να τονίσω τρία ζητήματα. Από μια πλευρά, ε, να ρωτήσω την Κομισιόν σε σχέση με την εξέλιξη των εμπορικών ροών εάν βασίζεστε στα στοιχεία της Eurostat ή της ε, Περιφερειακής Στατιστικής Υπηρεσίας της Κεντρικής Αμερικής, που σύμφωνα με εκείνη είναι ε, οι εξαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Κεντρική Αμερική αυξήθηκαν κατά 22% ενώ από την Κεντρική Αμερική προς την Ευρωπαϊκή Ένωση 17%. Σύμφωνα με τα ε, στοιχεία της Eurostat, η αύξηση των εμπορικών ροών ήταν αυξημένη εκτός από την Κωνσταντίνα. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν σε ποια στοιχεία αναφέρεστε και πού οφείλεται η διαφορά σε αυτά τα στοιχεία ανάμεσα Eurostat και Υπηρεσία Κεντρική Αμερική. Έπειτα υπάρχει πληροφορία για την, πληροφορίες για το εμπόριο υπηρεσιών. Έχουμε στοιχεία του 2014. Γιατί και μπορούμε να κάνουμε κάτι για να ε, βελτιώσουμε την ποιότητα των στατιστικών πληροφοριών ώστε να μπορούμε να έχουμε σωστά στοιχεία και να κάνουμε και εμείς σωστά τη δουλειά μας. Δεύτερον, όσον αφορά το μηχανισμό σταθεροποίησης για την μπανάνα, λειτουργήσε πολύ καλά. Δεν ξεπεράστηκαν τα όρια που θα έθεταν σε λειτουργία τις ε, ασφαλιστικές ε, δικλίδες, μόνο με τη Γουατεμάλα, λόγω του προβλήματος σταθεροποίησης της αγοράς και Ξέρετε πως υπάρχει μεγάλη ευαισθησία σε κάποια κράτη της Ένωσης όπου το εμπόριο της μπανάνας είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και είναι τόσο σημαντικός αυτός ο μηχανισμός σταθεροποίησης και ευτυχώς που λειτουργεί καλά. Τέλος, βιώσιμη ανάπτυξη. Όπως τόνισε ο εισηγητής, Έχουν γίνει ε, διάφορες συνεδριάσεις, όμως οι εκπρόσωποι της ε, κοινωνίας των πολιτών της Κεντρικής Αμερικής υπέβαλαν μια κοινή δήλωση και θέλω να γνωρίζω ποια ήταν η δική σας απάντηση από πλευρά της Κομισιόν. Και τι κάνει σε σχέση με το διάλογο ε, και το φόρουμ του διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών που από ό,τι ξέρω έγινε τον Ιούνιο του 2018 και πώς μπορούμε να δουλέψουμε για να ενισχύσουμε την κοινωνία των πολιτών και να βοηθήσουμε ώστε στην Κεντρική Αμερική να μπορέσουν να καταφέρουν τη δημοκρατία και τη βιώσιμη ανάπτυξη που χρειάζονται. Ευχαριστώ. Κύριος Γιώργενσον. Ευχαριστώ πολύ. Ε, νομίζω ότι η πολύ πλήρης ε, έκθεση διευκόλυνε πάρα πολύ το έργο μου γιατί ο εισηγητής συμπερέλαβε ορισμένα γενικά σημεία που, στα οποία ήθελα να αναφερθώ. Ε, συνολικά χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία αυτή από την πλευρά του Κοινοβουλίου. Είναι η κατάλληλη στιγμή ε, και θα γίνει και μια μελέτη εκτίμησης του αντεχτύπου αν όχι φέτος τον επόμενο χρόνο. Η συνολική μας αξιολόγηση είναι ότι είναι μια συμφωνία η οποία λειτουργήσε καλά στο σύνολό της και αν θέλουμε να εξετάσουμε τις ε, ροές αυτή τη στιγμή, έστω και αν το σύνολο του εμπορίου ε, δεν έχει αυξηθεί σημαντικά, μπορούμε παρόλα αυτά να διαπιστώσουμε ότι σε πολλούς ε, επιμέρους τομείς ε, το εμπόριο έχει αυξηθεί. Για παράδειγμα, από την Κωνσταντίνα κάποιον επιχειρήσεων που ασχολούνται με, με, με κομμάτια των υπολογιστών 45% ε, αύξηση ε, των εξαγωγών σε κάποιες από τις ε, περιοχές που ανέφερε και ο εισηγητής και αφορούν και ιατρικές συσκευές, καφέ κλπ. Όσον αφορά τις δικές μας εξαγωγές, πειράστηκαν από το γεγονός ότι υπήρξαν ε, πολλές ε, ε, καταγγελίες. μπορείτε να δείτε τους αριθμούς στον επόμενη έκθεση εφαρμογής που θα ακολουθήσει. Τώρα όσον αφορά τις, την ερώτηση που έθεσε η κυρία Πενιέρο όσον αφορά τους, ε, τα νούμερα. Πράγματι είναι πρόβλημα ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές ε, στους αριθμούς. Πιστεύουμε ότι ένας από τους λόγους θα μπορούσε να είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη ελεύθερη ζώνη εμπορίου στον Παναμά, η μεγαλύτερη στον κόσμο και τα στοιχεία της Eurostat ε, συμπεριλαμβάνουν αυτά τα στοιχεία, ενώ οι στατιστικές της ε, Κεντρικής Αμερικής περιλαμβάνουν μόνο τις ε, άμεσες εισαγωγές από τις δικές τους χώρες. Ε, εμείς θα συνεχίσουμε να βασόμαστε στα σχέδια της Eurostat. Χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα προτιμήσεων και θα πρέπει να συνεργαστούμε με την Κεντρική Αμερική γιατί δεν μπόρεσαν να μας παράσχουν τα στοιχεία αυτά. Σε σχέση με το Μεξικό, ε, δεν είναι μια υποχρέωση για αυτές τις ε, χώρες, ε, όπως για άλλους μας εταίρους, αλλά και ε, εδώ θα πρέπει να εργαστούμε τους ώστε να έχουμε στοιχεία. Όσον αφορά τις υπηρεσίες, είναι αλήθεια ότι ορισμένα από τα στοιχεία, την αριθμοί δεν είναι ακριβώ ενημερωμένοι, αλλά αυτό σχετίζεται ακριβώς με τη φύση των υπηρεσιών που υπάρχουν ε, αυτές οι καθυστερήσεις στα στοιχεία. Όπως είπατε, συμφωνούμε ότι το εμπόριο καθώς και η λειτουργία των θεσμών ε, έχουν λειτουργήσει σωστά όσον αφορά τις ε, ποστώσεις ανάκτησης. Εδώ μπορούμε να έχουμε κάποιες βελτιώσεις. Για τις μπανάνες η δική μας αξιολόγηση είναι το πλαίσιο είναι κατάλληλο. Θα πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα για την εφαρμογή. Χρειαζόμαστε πλήρη και σωστή εφαρμογή σε όλους τους τομείς και αυτό περιλαμβάνει και την βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που μας δίνει η συμφωνία ε, σε αυτούς τους τομείς, δηλαδή να επιστήσουμε την προσοχή αυτών των ε, χωρών στις υποχρεώσεις που έχουν όσον αφορά το εμπόριο και το περιβάλλον και να τις εφαρμόσουμε. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη δέσμευση και θα υποστηρίξουμε κάποια προγράμματα σε ολόκληρη την περιοχή αυτή και θα, αυτό συμπεριλαμβάνει και τη συνεργασία με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο πάνω μας εδώ εκπροσωπείται με την πρέσβυρα, στην οποία δίνω το λόγο για τέσσερα λεπτά. Με τον, τον κύριο πρέσβη. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Τέσσερα λεπτά είναι και υπερβολικά, γιατί ο κύριος Μπέγκε και ο κύριος Γιώργενσεν ήδη κάλυψαν τα όσα είχα να πω. Άρα η παρουσία μου εδώ είναι κάπως περίτη. Τέλος πάντων, νομίζω ότι μπορώ να επαναλάβω ότι πράγματι τα στοιχεία του εμπορίου για την ε, συμφωνία αυτή ε, σχηματίζουν μία εικόνα η οποία εκ πρώτης όψεως μοιάζει κάπως βαρετή αλλά εάν τα δείτε σε βάθος ε, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες ε, τις οποίες έχουμε εκμεταλλευτεί πέρα από αυτό οι ποσοστώσεις είναι ένα θέμα που σχετίζεται νομίζω εν μέρη με την ενημέρωση και τις συζητήσεις με τους εισαγωγείς και εξαγωγείς και κατά το οποίο ξέρω ότι οι συναδελφοί μου εδώ στις Βρυξέλλες και στην πρωτεύουσά μας ε, ε, είναι πολύ ευγνώμονες είναι τα ευρωπαϊκά προγράμματα που μας βοηθούν στην προώθηση της οικονομικής ολοκλήρωσης εντός του μπλοκ αυτού του οικονομικού για να μπορέσουμε ακριβώς να εκμεταλλευτούμε πλήρως την συμφωνία. Αυτό το οποίο μου απομένει να πω είναι ότι όπως είπε ήδη ο κύριος Μπέγκε είναι ότι εμείς θα θέλαμε να εφαρμοστεί πλήρως η συμφωνία αυτό σημαίνει ότι και, τα, και οι τέσσερις ή τρεις ε, εναπομείναντες εταίροι θα έπρεπε να κυρώσουν την συμφωνία το συντομότερο δυνατόν και υπ' την άποψη οτιδήποτε μπορούμε εμείς να κάνουμε για να βοηθήσουμε ε, ε, ευχαριστώ να το κάνουμε, να μιλήσουμε με τον κόσμο, με βουλευτές, με κλάδους που πιθανώς επηρεάζονται δουλειά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Κύριε Μπέγκε, ένα λεπτό για συμπεράσματα. Όχι, ωραία. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για το θέμα αυτό. Σημείο 22, διάφορα, το αγαπημένο μου, δεν υπάρχει τίποτα. Ωραία, η επόμενη συνεδρίαση 29 και 30 Αυγούστου και σας εύχομαι καλές διακοπές λίγη τη συνεδρίαση. Just after to see some of you, yes, people are you, just to talk about the composition of the